Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα για ψηφοφορία για, το, για την πρόταση αυτή τη και έτσι θα εγκριθεί όπως έχει. Προχωρούμε στη συζήτηση.